κυρίες και κύριοι συνεχίζουμε τη συνεδρίαση και σας καλωσορίζω θερμά για αυτήν την τελευταία ημέρα εργασιών της περίοδου συνόδου του Μαρτίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Αστρασβούργο. Τα πρακτικά των προηγούμενων συνεδριάσεων έχουν διανεμηθεί και ρωτώ αν υπάρχουν σχόλια. Όχι. Επομένως, θεωρείται ότι εγκρίθηκαν. Και πρώτο θέμα στην εμερική διάταξη. Έχουμε μία προφορική ερώτηση.